οποίος συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Ο κύριος Κρίστιαν Σίλβου Μπουσόη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ίσως θα πρέπει να διαλέξουμε με μια πιο καλή στιγμή μέσα στην εβδομάδα με μεγαλύτερη παρουσία βουλευτών. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση για πάρα πολλούς ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να βρούμε μια σαφή λύση για το μέλλον σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών. Ιδίω δεδομένου του γεγονότο ότι η δυνατότητα διαπραγμάτευση μεταξύ του καταναλωτή και τη ε, τράπεζα που δίνει το δάν, δάνειο είναι ανισομένη υπέρ τη τράπεζα. Δεν πρέπει λοιπόν να παρασυρθούμε από το λαϊκισμό, δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο το δοκιμαζόμενο τραπεζικό σύστημα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι αναλογική και εξισορροπημένη όπως λέει και ο κύριος Επίτροπος. Θα θέλαμε να ξέρουμε όμως ποια θα είναι η πρόταση αυτή της Κομισιόν για την επίτευξη λύσης. Μπορούμε να έχουμε την ε, λύση του λεγόμενου walk away, δηλαδή ότι τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να παραδώσουν το σπίτι τους και να μην έχουν καμία περαιτέρω ε, ευθύνη εναντί του Τραπεζικού Ιδρύματος. Δίνω τώρα το λόγο στον ε, κύριο Επίτροπο. τον Επιτρόπο Χίλ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, ήταν μια σύντομη συζήτηση σε μια χρονική στιγμή όταν δεν υπάρχει και μεγάλη προσέλευση βουλευτών. Λυπάμαι γι' αυτό γιατί το θέμα αυτό είναι παρόλα αυτά εξαιρετικά σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ίσως το πιο σημαντικό σημείο εκκίνησης είναι τι πρέπει να πράξουμε για να προστατεύσουμε στο μέλλον τους καταναλωτές. Όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, εξαρτάται από την νομοθεσία για τα στεγαστικά δάνεια που θα δημιουργήσει ένα καλύτερο πλαίσιο με πιο ε, αποτελεσματικές θεραπείες για να προστατεύσουν τους καταναλωτές όταν υπάρχει σημαντική αλλαγή ισοτιμιών και αυξηθεί, το κόστος εξυπηρέτησης του στεγαστικού δανείου. Πιο γενικά όμως αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις ε, υπηρεσίες για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια χρειάζεται να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία και ποιότητα στην αγορά ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να διαλέγουν με καλύτερα. Γιατί αν δείτε, όπως είπε και ο κύριος Κέλλη, την ε, τιμολόγηση ορισμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποικίλει πάρα πολύ η τιμολόγησή τους. Και μία από τις ιδέες ε, μέσα στην πρόταση για την ε, ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι να ενισχύσουμε για για λιανοπολικές ε, υπηρεσίες, για απλούς καταναλωτές να ε, εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ομοιογένεια σε αυτήν την αγορά, όχι προς όφελος των μεγάλων χρηματοπιστωτικών φορέων, αλλά των απλών πολιτών. Ξεκινώ λοιπόν με αυτό, γιατί η σημασία του να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια πιο στεναρή ε, ενιαία αγορά για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συνδέεται με την ανάγκη να υπάρχουν ελεύθερες ροές κεφαλαίων και ενιαία κεφαλαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπανε πολλοί συνάδελφοι. Και αυτό είναι και η προσέγγιση που έχει ακολουθήσει η Κομισιόν στην περίπτωση των δανείων σε ξένα νομίσματα. Όπω είπαν πολλοί συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ξεβρούμε μια ισορροπία, μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των καταναλωτών αφενό και των τραπεζικών φορέων. Και προφανώ από την οπτική αυτή γωνία των καταναλωτών πρέπει τα κρατημέλη να προστατεύσουν τους καταναλωτές. Είναι απόλυτα θεμητό. Αν θέλουμε όμως συγχρόνως να διατηρήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ενιαία αγορά κεφαλαίων θα πρέπει να έχουμε και ένα νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι χρηματοπιστωτικοί φορείς και να εξασφαλίσουμε ότι όταν οι κυβερνήσεις παίρνουν τέτοιες κάνουν τέτοια μέτρα για να προστατεύσουν τους καταναλωτές, το κάνουν μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά ε, βρίσκονται στη βάση της προσέγγισης που η Κομισιόν προσπαθεί να αναπτύξει μαζί με ορισμένα κράτη-μέλη. Απαντώντας σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, με ρωτήσανε πόσα κράτη-μέλη ε, διαβουλεύτηκαν ε, εκ των προτέρων με την Κομισιόν προτού πάρουν μέτρα. Τα κράτη-μέλη βέβαια δεν είναι υποχρεωμένα να συμβουλευτούν την Κομισιόν προτού <clears throat> νομοθετήσουν στα θέματα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Εμεί εποπτεύουμε τα μέτρα αυτά στη Ρουμανία και την Πολωνία, γιατί εκεί τα κράτη-μέλη μα έχουν δώσει τη, τα σχέδια νόμου για τα θέματα αυτά και συζητούμε επίσης με την κυβέρνηση της Κροατίας για να δούμε αν μπορούμε να εξεύρουμε μια αξισορροπημένη λύση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτό όπως ελέγχθη, μάλλον όπως ελέγχθη δεν ισχύει το ότι η Κομισιόν έχει σαν στόχο να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά χωρών οι οποίες πήραν τέτοια μέτρα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ τόνισα προηγουμένω ότι είναι απόλυτα θεμητό για τι κυβερνήσει να αναλαμβάνουν τέτοιε ενέργειε, τέτοιε δράσει, αλλά όπω είπαν πολλοί συνάδελφοι, το θέμα τη αναδρομικότητα των αποφάσεων αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Το θέμα τη αναλογικότητα επίση έχει μεγάλη σημασία. Και το να μην υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των κυβερνήσεων στην ομοθεσία τους μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών καταναλωτών, αυτό είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να εξεύρουμε μια πρακτική ρύθμιση για όλα αυτά τα προβλήματα και εγώ ενθαρρύνομαι από την υποστήριξη που πήρα από ένα αριθμό μέλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσωπικά θα συνεχίσω να είμαι προσιλωμένο στη συνέχεια αυτού του έργου, θα είμαι σε επαφή με τους αρμόδιους υπουργού και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την απαιτούμενη πρόοδο για να μπορέσουμε να δώσουμε σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αλλά συγχρόνως και προστασία για του καταναλωτέ. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την Κροατία, εμείς συνεχίζουμε την αξιολόγηση της κατάστασης για να εξασφαλίσουμε το ότι οι ενέργειες που γίνονται από την κροατική κυβέρνηση συνάδουν με την ενιαία αγορά και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κροατία βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Θα εξακολουθήσουμε να ασκούμε πίεση και παρακολουθούμε και τα τεκτενόμενα σε άλλες χώρες όπου μπορούν να ληφθούν και εκεί μέτρα σε σχέση με τα δάνεια σε ξενονόμισμα για να ελέγξουμε ότι πράγματι συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι σημαντικό όμως το θέμα αυτό θα το έχουμε πάντα μπροστά στα μάτια μας και να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει προστασία των καταναλωτών, αλλά συγχρόνως υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο και σεβόμαστε το κράτος δικαίου. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν με <clears throat> βεβαιότητα, γιατί αν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις και να έχουμε μια ένωση κεφαλαίου αγορών, χρειάζονται οι επιχειρήσεις να ξέρουν ότι έχουν μια βεβαιότητα και μπορούν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την τόσο σημαντική αυτήν δήλωση και με τον τρόπο αυτό κλείνει η συζήτησή μας.